Dear um, Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε. Δεν θέλω να ε, ζωρίσω το χρόνο σε, για αυτή την πολύ σημαντική παρουσίαση. Αν θέλουμε, ας ξεκινήσουμε μια σημαντική ομιλία από τον Μάικλ Φλάιρτη. Καλώς όρισες, ε, Μάικλ. Χαίρομαι που σε καλωσορίζω. Είσαι ο Διευθυντής του ε, Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παρουσιάσεις το ετήσιο πρόγραμμα και τις προτεραιότητες για το 2018. Οι συνάδελφοι γνωρίζουν, αλλά καλό είναι να επαναλάβουμε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τεκμηριωμένες πληροφορίες και δεδομένα και βοήθεια στον τομέα των, ε, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολλοί τομείς στους οποίους ο οργανισμός έχει αναπτύξει τη δουλειά του τα τελευταία χρόνια σε θεματικούς τομείς που αφορούν και το ε, πολιετές πλαίσιο. Θέλω να <clears throat> ευχαριστήσω τον οργανισμό δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Μάικλ θα αναφερθεί ε, στα θέματα αυτά, αλλά θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί, ε, ευχαριστήσω γιατί μας έφερε πιο κοντά. Ένα από τα βασικά θέματα για την επίσκεψη που έγινε, θέλω να αναφερθώ στο θέμα των, της ε, βοήθειας που προσφέρει ο οργανισμός σε κράτη-μέλη και αυτό είναι ένα θέμα που έχει τεθεί, όπως επίσης και πολλά άλλα διαρθρωτικά και στρατηγικής φύσεως θέματα που θα θα θίξει ο Μάικλ και την πρόοδο που είναι προφανής και την οποία θα θέσει, θα παρουσιάσει. Έχουμε πλέον λάβει την ανεξάρτητη αξιολόγηση του οργανισμού με βάση το άρθρο 31 του κανονισμού του και υπάρχει στην ιστοσελίδα. Άρα θα ζητήσω από τον Μάικλ κατευθείαν να κάνει την παρουσίασή του για το 2018, δηλαδή το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του οργανισμού για 12-13 λεπτά και μετά θα αρχίσει η συζήτηση. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς και τα αξιότιμα μέλη για την πρόσκληση. Θέλω να σας ευχαριστήσω και προσωπικά που ήρθατε και μας επισκεφτήκατε. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, κυρίως και για να, καταλάβετε καλύτερα τις για να καταλάβουμε καλύτερα τις προτεραιότητες της Επιτροπής και να ε, κινηθούμε ανάλογα. Αξιότιμα μέλη δεν ε, μπαίνω στο 2018 με μεγάλη αισιοδοξία. Δεν πιστεύω ότι η κατάσταση θα είναι πολύ καλύτερη από το 2017 που ήταν μια ε, χρονιά γεμάτη προκλήσεις. Βλέπουμε μορφές ε, βίας που είναι απαράδεκτες, πάρα πολλές παραβιάσεις από πολλούς ηγέτες σε πολλά μέρη και επίσης την πεποίθηση του γενικού πληθυσμού ότι τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα τους αφορούν και ότι έχουν σημασία. Παρά τις ε, για να αλλάξουν αυτές οι τάσεις πρέπει όλοι να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβουμε ηγετική θέση στο σύνολο αυτής της προσπάθειας. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα συνεχίσει να στηρίζει τον ηγετικό σας ρόλο για την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής. Για να υποστηρίξουμε εσάς και τα άλλα θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο μας ε, το Δεκέμβριο πέρυσι ενέκρινε ένα πενταετές στρατηγικό σχέδιο που λαμβάνει υπόψη το πολιετές σχέδιο, το θεματικό πλαίσιο που συμφώνησαν οι, τα θεσμικά όργανα για μας, όπως επίσης και την ανεξάρτητη αξιολόγηση που ανέφερε μόλις τώρα ο Πρόεδρος. Φυσικά κάθε χρόνο <clears throat> έχουμε ετήσια προγράμματα εργασίας. Το πρόγραμμα εργασίας του 2018 περιλαμβάνει 45 ε, χωριστά έργα. Δεν θα τα αναφέρω όλα αυτά, κάποια μόνο, τα οποία ενδεχομένως σα ενδιαφέρουν περισσότερο ως Επιτροπή. Πρώτον, πριν από λίγες μόλις εβδομάδες ε, δημοσιεύσαμε μια έκθεση που ήταν η χρονιά εν το για το θέμα του χώρου της κοινωνίας των πολιτών εντός της Ένωσης. Θεωρούμε ότι και στα 28 κράτη-μέλη υφίστανται πιέσεις με πολλές διαφορετικές μορφές. Το θέμα όμως είναι ότι οι πιέσεις στην κοινωνία των πολιτών είναι τόσο στο, υπάρχουν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Ένωσης. Ξεκινήσαμε το έργο αυτό με βάση του ιδρυτικού μας κανονισμού, ο οποίος ζητά να συνεργαζόμαστε στενά με την κοινωνία των πολιτών. Άρα έχουμε οριζόντια ευθύνη να ελέγξουμε την κατάσταση υγείας και να στηρίξουμε ε, την, ε, την ευημερία και την καλή κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα κράτη-μέλη. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πιέσεις στα κράτη-μέλη και οικονομικών πιέσεων και θεσμικών και δυστυχώς σε πολλά μέρη με τη μορφή ομών ε, απειλών σε άτομα και ε, περιουσίες. Βεβαίως βρήκαμε και καλές πρακτικές σε κάποια κράτη-μέλη, οποία, τις οποίες πρέπει να προσέξουμε. Η έκθεση ολοκληρώθηκε με κάποιες συστάσεις για θέματα όπως η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, η φροντίδα με τους οποίους πρέπει να ε, συντάσσονται οι νόμοι που αφορούν και η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρακολουθεί τις μορφές πίεσης επί της κοινωνίας των πολιτών όπως ε, εμφανίζονται. Φυσικά όλο το χρόνο θα συνεχίσουμε το έργο αυτό. Ένας δεύτερος τομέας ε, εργασίας ε, που θα αναφέρω ως παράδειγμα είναι το θέμα των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων που προκύπτουν με τον, για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μεγάλης κλίμακας συστήματα πληροφορικής. Το έργο μας αφορά εννέα εκρεμείς ε, νομοθετικούς φακέλους και βάσει αυτής της δουλειάς έχουμε εκδώσει ε, τρεις νομικές, τρεις νομικές γνωμοδοτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο σχετικός φάκελος θα δημοσιευθεί στις 28 Μαρτίου. Θα ήθελα να αναφέρω από τώρα κάποια βασικά θέματα θεμελιδών δικαιωμάτων που εντοπίσαμε στην έρευνα που έχουμε κάνει εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Πρώτον, υπάρχει ένα θέμα των αυτών οι οποίοι υπόκεινται στη συγκέντρωση δεδομένων, που οι οποίοι δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους όσον αφορά τα δεδομένα αυτά που τους αφορούν, αυτούς και τις δραστηριότητές τους. Δεύτερον, μας ανησυχεί το θέμα της ακρίβειας των δεδομένων στο πλαίσιο αυτών των συστημάτων, διότι ένα σφάλμα σε ένα σύστημα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ε, ανησυχίες στον τομέα των θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό μας οδηγεί σε έναν άλλο δύσκολο χώρο που de facto αφορά το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτούς που υπόκεινται στη συγκέντρωση στοιχείων ε, για, ε, για διόρθωση των στοιχείων των λάθων που έχουν ήδη εισαχθεί. Επίσης, το θέμα της διαλειτουργικότητας των μεγάλων αυτών συστημάτων έχουμε δημοσιεύσει μια ειδική έκθεση στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στην, ε, στην ομάδα υψηλού επίπεδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί αναφέρουμε σχεδόν όλα όσα είπα τώρα και πολλά άλλα και στο συγκεκριμένο ε, θέμα της διαλειτουργικότητας επικεντρωνόμαστε στο θέμα του να τηρείται η αρχή της, του περιορισμού με βάση το σκοπό η έρευνα έχει δείξει ότι η διαλειτουργικότητα δεν είναι απλώς δύσκολη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά μπορεί να δώσει και πολύ θετικά αποτελέσματα όσον αφορά παραδείγματος χάρη την παρακολούθηση, τον εντοπισμό παιδιών που έχουν χαθεί. Ε, υπάρχουν προτάσεις ενώπιών σας αυτή τη στιγμή και θεωρούμε ότι έχουμε ευρήματα που έχουν σχέση με αυτά που θα συζητήσετε. Όμως θέλω να επισημάνω ότι κάποια στοιχεία των προτάσεων που μελετάτε δεν τα μελετήσαμε γιατί δεν εμπίπτουν στις συζητήσεις ε, της ομάδας ψηλού επίπεδου. Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που αφορούν την ε, αυτούς, ε, τις συσκευές που εντοπίζουν πολλαπλές ταυτότητες και το αποθετήριο κοινή ταυτότητας. Θα θέλαμε το Κοινοβούλιο να ζητήσει νομική γνωμοδότηση για το θέμα της διαλειτουργικότητας από τον οργανισμό και με τα χαρά θα την παραδώσουμε. Επίσης, θέλω να προτείνω στην Επιτροπή, αν σας ενδιαφέρει, θα ήταν θετικό για μας να σας παρουσιάσουμε λεπτομερέστερα τα, ευρήματα, τα ευρήματα της έρευνάς μας στον τομέα των βιομετρικών δεδομένων. Τώρα, το θέμα της δουλειάς που κάνουμε στα ε, κέντρα συγκέντρωσης των μεταναστών, τα hot spots, είναι μια δουλειά που συνεχίζεται εδώ και δύο χρόνια και πριν από λίγες εβδομάδες υπογράψαμε μια ένα νέο μνημόνιο ε, συνεννόησης με την ελληνική κυβέρνηση για την παράταση της συνεργασίας κατά ένα χρόνο. Τι κάνουμε. Στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, μας παρακολουθούμε σωστά τις, διαδικα... τις μόνιμες διαδικασίες λειτουργίας ε, των κέντρων συγκέντρωσης και φιλοξενίας για να εξασφαλίσουμε ότι συνάδουν με την νομοθεσία στον τομέα παραδείγματος χάρη προστασίας των παιδιών. Επίσης υποστηρίζουμε την ελληνική κυβέρνηση η οποία επιδιώκει να αναθεωρήσει τα θέματα κυδαιμονίας. Τώρα όσον αφορά την Ελλάδα ένα θέμα που μας ανησυχεί τώρα είναι το θέμα της βίας ε, ε, ε, σεξουαλικής και με βάση το φύλλο. Θέλουμε να χαρτογραφήσουμε τις δυνατότητες να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό σε όλα τα κέντρα στα ελληνικά νησιά. Όσον αφορά τώρα την εμπλοκή μας με τα hot spot, πρόσφατα γιορτάσαμε τη δεύτερη επέσιο της ε, υποβολής έκθεσης κάθε μήνα. Κάθε μήνα, τα τελευταία δύο χρόνια, υποβάλλουμε μια λεπτομερή έκθεση με δεδομένα όχι στα ε, όλα τα hot spot, αλλά στα ε, κράτη-μέλη που επηρεάζονται περισσότερο. Και σε μια συνολική έκθεση πριν από λίγες εβδομάδες μπορέσαμε να εντοπίσουμε πέντε τομείς που διαρκώς δημιουργούν προβλήματα στα 14 κράτη-μέλη που παρακολουθούμε όπου κάνουμε αυτή την ανάλυση. Καταρχήν, είδαμε ότι υπάρχουν μόνιμες δυσκολίες πρόσβασης στις διαδικασίες αιτήσεως ασύλου. Δηλαδή, η πρόσβαση είναι πιο περιορισμένη σε κάποια κράτη-μέλη από ό,τι πριν από δύο χρόνια. Δεύτερον, από την ώρα που υπάρχει αυτή η πρόσβαση στις διαδικασίες υποβολής αιτήσεως ασύλου, ε, συνήθως είναι πολύ χρονοβόρα και οι ίδιες οι διαδικασίες μερικές φορές είναι προβληματικές όσον αφορά ας πούμε το δικαίωμα υποβολής ε, έφεσης. Δεύτερον, ε, κατόπιν εξακολουθούμε να βλέπουμε προβλήματα στις εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται οι μετανάστες και αυτό με ανησυχεί πολύ ε, γιατί μιλάμε για το, μέσο του χειμώνα και μια βασική, ένα βασική να υπάρχει μια στέγη και λίγη θέρμανση. Και αυτό γίνεται σε πολλά μέρη. Τέταρτον, το θέμα της προστασίας των παιδιών εξακολουθεί να παραμένει ανησυχητικό όπως και τα τελευταία δύο χρόνια. Και τέλος, ανησυχούμε από την υπερβολική πρόσβαση στην κράτηση των μεταναστών συμπεριλαμβανομένων και των, ποδιών, ε, των παιδιών εντός των διαδικασιών. Τα, τα κέντρα κράτησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως τελευταία λύση. Αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να έχουμε μια συγκεκριμένη ανταλλαγή απόψεων με πολύ πολύ περισσότερες λεπτομέρειες σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχουν σχέση με την κατάσταση του μεταναστευτικού και κάτι ευρύτερο από ότι τη, απλώς η κατάσταση στα hot spot. Τώρα, ένα άλλο θέμα, τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ρωμά. Ε, θα ε, δημοσιεύσουμε το 2018 δύο... Ε, ε, ε, θα κάνουμε δύο δημοσιεύσεις τον Απρίλιο το πρώτο που θα είναι οι, οι ε, για την ε, στροφή κατά των τσιγκάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και αυτό στηρίζεται στην δουλειά η ευρωπαϊκή Ένωσης ΜΑΙΔΑΣ που θα, και το, σχέδιο, το προσχέδιο είναι σχεδόν έτοιμο. Δεύτερον, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να απομονώσουμε το θέμα του φύλου από τη δουλειά μας όπου είναι δυνατόν και το Σεπτέμβριο θα κάνουμε μια τέτοια δημοσίευση για την συγκεκριμένη εμπειρία των διακρίσεων για γυναίκες και ε, Ρωμά και μετανάστριες. Αυτό θεωρούμε ότι θα βοηθήσει πολύ στην καλύτερη κατανόηση ε, της κατάστασης και της συγκεκριμένη εμπειρίας που ζουν οι γυναίκες Ρωμά σε σχέση με τους άνδρες που υφίστανται μεγάλες διακρίσεις και ε, διώξεις. Τώρα, στο κράτος δικαίου το θέμα της προστασίας και υποστήριξης του κράτους δικαίου είναι πολύ ευρύτερο από τα θεμελιώδη δικαιώματα, πολύ ευρύτερο από την εντολή που έχει ο οργανισμός μας. Όμως τα, ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα έχουν μεγάλη σχέση της σημασίας της στήριξης του κράτους δικαίου και σκοπεύουμε να προσφέρουμε κάθε δυνατή υποστήριξη στο πλαίσιο αυτό. Μια από τις σημαντικότερες προσφορές μας το 2018 θα είναι η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα. Ένα σύστημα όπου όλα τα ευρήματα που αφορούν κάθε κράτος μέλος, ε, όλα τα δικαστικά και τα ε, σχετικά ευρήματα θα μπορούν να αναζητηθούν αναχώρα και κατηγορία. Και πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να στηρίξουμε τη δουλειά σας. Ένα τελευταίο τομέα εργασία μα είναι ότι το 2018 σημειώνονται δύο χρόνια από το 2016 όπου έγινε το πρώτο φόρουμ του θεμελιωδών δικαιωμάτων. Που σημαίνει ότι είναι κατάλληλη στιγμή να γίνει το δεύτερο φόρουμ που θα γίνει από τι 25 27 Σεπτεμβρίου στη Βιέννη. Θα αποτελέσει σημαντική πρωτοβουλία για να ξεκινήσουν διαφορετικές συζητήσεις και ε, περισυλλογή ε, μεταξύ ανθρώπων που δεν συναντώνται συνήθως για να πορευτούν στο δρόμο της ισχυρότερης προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης. Τώρα το ε, βασικό θέμα θα είναι το ανήκει, δηλαδή πώς θα τους φέρουμε όλους μέσα στην σκηνή μας και από την ώρα που θα έρθουν εκεί πώς θα τους φερθούμε με σεβασμό με βάση την πολυμορφία τέτοιου είδους συναντήσεις, συζητήσεις δεν γίνονται. Θα ακούσουμε ε, ψηλά στελέχη του ε, Ηνωμένων Εθνών, τη Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ανθρώπους από την κοινωνία των, ε, πολιτών. Θα έχουμε ομάδες θρησκευτικέ, άλλες κοινότητες και θα το οργανώσουμε με πολύ φαντασία. Ε, που θα δώσει, πράγμα θα δώσει καλά αποτελέσματα. Την προηγούμενη φορά υπήρχε μια εντυπωσιακά ισχυρή και δημιουργική ε, αντιπροσωπεία της Επιτροπής σας και προσβλέπουμε ε, στο να συμμετάσχετε και να εμπλουτίσετε στις συζητήσεις όπως πράξατε και το 2016. Βεβαίως την κατάλληλη στιγμή θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας για τα ε, συνέχεια που θα δοθεί στα αποτελέσματα του φόρουμ. Και κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα δύο λόγια να πω για τα θεσμικά θέματα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Όπως γνωρίζετε, είχαμε την εμπειρία εξωτερική αξιολόγηση του οργανισμού που είδε τις επιδόσεις μας σε πέντε τομεί, που, πόση σημασία έχουμε, πόση αποτελεσματικότητα έχουμε, πόση προστιθέμενη αξία προσφέρουμε, τι συντονισμό γίνεται και τι αποτελεσμα, πόσο αποτελεσματικοί είμαστε. Και πρέπει να πω ότι είχαμε καλή βαθμολογία σε όλους αυτούς τους ε, τομείς. Η αξιολόγηση οδήγησε σε κάποιες συστάσεις για το πώς θα κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας τις οποίες μελέτησε το Δεκέμβριο το Διοικητικό Συμβούλιο. Και τώρα θα σας παρουσιάσω παρότι θα σας αποσταλεί επισήμως, θα σας παρουσιάσω κάποιες από τις συστάσεις που ε, ε, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα σας, ε, τρία, θα σας δώσω τρία συμπεράσματα, κανένα από αυτά δεν θα σας εκπλήξει. Πρώτον, το, το γεγονός ότι ο οργανισμός δεν έχει σαφή εντολή να κινηθεί από μόνη της σε θέματα αστυνομικής και δικαστική συνεργασία σε ποινικών θεμάτων. Έτσι ζητάμε να μα δοθεί ε, ρητή εντολή σε αυτό το τομέα, ρητή δικαιοδοσία. Δεύτερον, ε, συνιστά το Διοικητικό Συμβούλιο να μα δοθεί η δυνατότητα να γνωμοδοτούμε επί σχεδίων ε, νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδία πρωτοβουλία. Όπω είπα προηγουμένω, μπορούμε να λειτουργήσουμε επί τέτοιων θεμάτων μόνο μετά από αίτημα ενό θεσμικού οργάνου που συνήθως είναι το Κοινοβούλιο. Και τρίτον και τελευταίο, το Διοικητικό Συμβούλιο επεσήμανε ότι δεν έχουμε επαρκείς πόρους. Δεν μπορούμε να πετύχουμε ούτε κατά διάνοια αυτά τα οποία ε, πρέπει να πετύχουμε με τους περιορισμένους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, ε, εν κατακλείδη θέλω να υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή αυτή ε, γνωμοδοτεί όσον αφορά την, ε, τον διορισμό της επιστημονικής μας επιτροπής. Είναι ένα θέμα που για μας είναι πολύ σοβαρό. Η ανεξάρτητη επιστημονική ε, ε, επιτροπή μας είναι μία από τις θετικές πρακτικές του οργανισμού που εξασφαλίζει ότι τα αποτέλεσμα των ερευνών μας είναι υψηλωτά του επίπεδου. Θα θέλαμε λοιπόν να σας ζητήσουμε να μελετήσετε πολύ προσεκτικά τον κατάλογο που έχετε ενώπιόν σας, να βοηθήσετε το Δικικό Συμβούλιο να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Και τέλος, σύντομα θα έρθει η Αυστριακή Προεδρία, πράγμα που πιστεύω θα προσφέρει πολλές ευκαιρίες ε, σε εσά να επισκεφτείτε τη Βιέννη. Και πέρα από το Φόρουμ Θερμιλωδών Δικαιωμάτων θα ήθελα να προσκαλέσω όποιον θέλει, όποιο μέλος Επιτροπής σας θέλει να μας επισκεφτεί στον οργανισμό, να επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις μας για να καταλάβετε καλύτερα τι κάνουμε αυτή την εποχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Μάικλ. Μερικά σημεία να τονίσω κι εγώ. Πρώτον, βεβαίω θα συμμετέχουμε απολύτω και πλήρω στο φόρουμ αυτό και σα ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω μερικά πράγματα. Ε, πρόσφατα μετέβηνε στη Βιέννη και είδα και το Διευθυντή και το Προσωπικό και το ε, Διοικητικό Συμβούλιο και είχαμε αρκετά εντατικές συζητήσεις και τονίσατε και εσείς τα ίδια θέματα που είπατε και εδώ. Μπορεί να θέλουν οι συνάδελφοι να σχολιάσουν αυτά που ακούσατε για τις πρωτοβουλίες ε, γνωμοδότης. Μιλήσατε για τους πόρους, την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ε, ποινικά θέματα. Τα σημειώσαμε όλα αυτά και είχα πει ότι θα τα θέσω και υπόψη της Επιτροπής μας, τα κάνατε κι εσείς. Είναι προφανές ότι καλύπτεται μια τεράστια ε, περιοχή, τομέα αρμοδιοτήτων από πλευράς πολιτικής, αλλά υπάρχουν και κάποια πρακτικά ζητήματα. Κάνετε πάρα πολλές εκθέσεις και αυτό το είδαν και άλλοι συνάδελφοι που πήγαν στη Βιέννη. Είναι πανεπιστημιακού επίπεδου αυτή η δουλειά που κάνετε και μπορούν και μεμονωμένοι βουλευτές να προσφύγουν σε εσά. Και μάλλον δεν το γνωρίζουν πολύ καλά, ή δεν το έχουν ε, χωνέψει. Δεν είναι μόνο τα θεσμικά όργανα, μπορούν και οι βουλευτές να ζητήσουν τη βοήθεια του οργανισμού της Βιέννης. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να ανταποκριθεί ο οργανισμός σε αυτό το πεδίο που έχει τόσο εντατική ε, δουλειά αυτό τον καιρό χωρίς ε, άμεση διαπροσωπική επαφή, εισηγητέ, διάφοροι ενδιαφερόμενοι, να το έχετε υπόψη σας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αρχίζει η συζήτηση. Θα δώσουμε πρώτα το λόγο στην κυρία Κινίτση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ ε, και τον Διευθυντή, τον κύριο Μάικλ ο Φλάχερτη που μας παρουσίασε τις μεγάλες προκλήσεις που μας περιμένουν και το 2018 ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, ακούσαμε να μας αναλύεται πολλά σημεία και θέλω να συγχαρώ τον οργανισμό για το έργο του αλλά και τη συνεισφορά του στις δικές μας εργασίες. Σήμερα οι προκλήσεις εξακολουθούν να είναι πολλαπλές, δυστυχώς, τρομοκρατία, μεταναστευτική κρίση και πάει λέγοντας. και είναι πολλές οι απειλές για τα θεμελιώδη δικαιώματα και μέσω του διαδικτύου. Και νομίζω ότι αυτού του είδους η έρευνα είναι πάρα πολύ σημαντική και συγκεκριμένα η προστασία των ανηλίκων. Ε, το ίντερνετ και τα ε, κοινωνικά δίκτυα ε, είναι μια πλατφόρμα γνώσης, ανταλλαγής επικοινωνίας, ε, και χρησιμοποιείται από όλο και νεότερους πλέον ανηλίκους. Αλλά υπάρχουν κίνδυνοι, τα γνωρίζετε, και εξτρεμισμού και εγκλημάτων, μαστροπίας κλπ. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω κάτι για το μέλλον. Ποιες είναι οι δυνατότητες που διαθέτουμε έτσι ώστε να ε, επικεντρώσουμε και να εστιάσουμε τη δική μας προσοχή εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προστασία των ανηλίκων απέναντι σε αυτούς τους διαδικτυακούς κινδύνους. Εσείς ε, μιλήσατε για πολλά θέματα, αλλά για τους ανηλίκους επίσης, για να παραμείνω σε αυτούς, ε, η κράτηση παιδιών είναι κάτι ε, τέλειως απαράδεκτο. Πέρσι, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επίτροπη Γιούρη Νομικών ε, Θεμάτων ασχολήθηκε με το θέμα αυτό της κράτησης των ανηλίκων. Για να τερματιστούν αυτά τα φαινόμενα και να μπορούν οι ανήλικοι να χαίρουν προστασίας. Ένα άλλο θέμα είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι και η προστασία τους. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ποια είναι η θέση του οργανισμού σας ως προς την αναθεώρηση του κειμένου Eurodac, όπου τώρα προβλέπεται ταυτοποίηση ανηλίκων, οι οποίοι όμως χρειάζονται προστασία, ιδιαίτερα συνόδευτοι. Όταν είναι γνωστή η ταυτότητά τους, για να μπορούμε να παρακολουθούμε τις μετακινήσεις τους. Αυτό το κείμενο ακόμα δεν έχει συμφωνηθεί, είναι στη συζήτηση. Και μιλούν για δακτυλικά αποτυπώματα που θα παίρνουν από παιδιά μέχρι ηλικία 6 ετών. Από 6 ετών και πάνω. Και πώς θα γίνει αυτό. Και μπορεί να γίνει χρήση βίας Γιατί τη δακτυλοσκόπηση των πιο μεγάλων ε, ανηλίκων που δεν είναι παιδιά αλλά παραμένουν ανήλικοι. Είναι 17 ετών ας πούμε. Ε, δεν θα μακρηγορήσω γιατί θέλω να μιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι. Αναφερθήκατε και σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που είναι οι εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις που υφίσταται η κοινωνία μας. Αυτό μου θύμισε το εξή πολύ σημαντικό που συνδέεται και με την τρομοκρατία. Γνωρίσαμε ένα, ένα κύμα συγγνώμη, τρομοκρατίας που οδήγησε σε διακρίσεις σε κάποιες χώρες απέναντι στη μουσουλμανική κοινότητα με όλα τα συμπαραμαρτούντα. Και ασκούνται μεγάλες πιέσεις στην κοινωνία που μπορούν να επιφέρουν επεισόδια διακρίσεις εις βάρος της κοινότητας και αντιδράσεις ε, από πλευράς εκείνων που δεν αισθάνονται ευπρόσδεκτοι ούτε ενταγμένοι στην κοινωνία, ενώ θέλουν να ενταχθούν και να συμμετέχουν. Αυτά ήθελα να σας αναφέρω και θα παρακαλούσα να μας απαντήσετε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόνι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ ε, για την παρουσίαση αυτή την τόσο εμπεριστατωμένη και εξαντλητική για το 2018 και τις προτεραιότητες που είναι πάρα πολύ χρήσιμες και, και εύστοχα αυτά που λέτε. για μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, βεβαίως, οι μετανάστες, τα hot spots ε, ε, είναι σημαντικά θέματα, ο αντιτσιγκανισμός, αλλά επίσης θα πρέπει να παρακολουθούμε και κάποια νέα φαινόμενα. Δυστυχώς ε, είναι φαινόμενα αντισημιτισμού που αναδύονται και είναι πραγματικό πρόβλημα αυτό στις ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης και φυσικά όταν μιλούμε για το κράτος δικαίου έχει μεγάλη σημασία να μην αναφέρουμε μόνο κάποια συστήματα, το δικαστικό σύστημα, το πρόβλημα κάποιο σύστημα στην Πολωνία ας πούμε, αλλά να δούμε τι αποτελέσματα επιφέρουν ε, στην ε, καθημερινή ζωή των πολιτών, των ανθρώπων αυτές οι αλλαγές και οι ε, μεταρρυθμίσεις. Χρειάζεται παρακολούθηση η κατάσταση. Δηλαδή, απειλείται πραγματικά η ζωή των πολιτών ή όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί οι εκθέσεις σας ε, θα ασχοληθούν και με θέματα ψηφιακά, ε, ζητήματα δεδομένων, ακρίβεια των δεδομένων, πρόσβαση στα δεδομένα και όλα αυτά. Δυνατότητα διόρθωσης ακόμα και ε, απάλληψης κάποιων. Και επειδή έχουμε την εφαρμογή του GDPR, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και τη ε, ιδιωτική σφαίρα. Ένα τελευταίο έχει να κάνει με την έκθεση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκθέση. Αυτή είναι εξαιρετική, το τονίζω, εξαιρετική και χρειάζεται και συζήτηση για πολλά θέματα που άπτονται της έκθεσης. Είναι μια πρόταση προς τον Πρόεδρο και προς εσάς αυτή, γιατί ο οργανισμός σας έχει καταθέσει, έχει παρουσιάσει εννέα γνωμοδοτήσεις. Ουσιαστικά συστάσεις είναι αυτές. Και νομίζω ότι θα πρέπει καμιά φορά να επανερχόμαστε στις συστάσεις σας αυτές. Όχι να έχουμε την έκθεση απλώς, αλλά να δίνουμε και συνέχεια. Να δημιουργούμε μια κατάσταση όπου θα μπορούμε να αντιδρούμε σε αυτές τις ε, προτάσεις και τις νομοδοτήσεις και τις συστάσεις σας, ας πούμε. Ανεξάρτητη χρηματοδότηση της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό είναι ένα θέμα που θα βρούμε μπροστά μας όταν θα καταρτήσουμε το ψήφισμα για τη χρηματοδότηση με ανεξάρτητο τρόπο των οργανώσεων που ασχολούνται με την οικοδόμηση δημοκρατίας, κράτους δικαίου και της κοινωνίας ε, που να αντιλαμβάνεται την ηθαγένεια. Ε, ευχαριστώ κύριε Μπόνη. Αυτό το θέμα είναι σε πολλές συστάσεις και γνωμοδοτήσεις, πραγματικά πολύτιμη δουλειά και έρευνα και τα χρησιμοποιούμε. Αλλά πώς τα χρησιμοποιούμε είναι ένα άλλο θέμα. Χρειάζεται βελτίωση. Γιατί το περιεχόμενο αυτό πραγματικά μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο. Και η γνωμοδότηση για τη Eurodac ε, επίσης ε, μιλάει για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους του οργανισμού ΦΡΑ. Και είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίασή σας και σε αυτήν μας είπατε ότι στην κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη περνάμε μια κρίση. Ε, και εκεί πραγματικά σε αυτό το επίπεδο βρίσκεται και η ευθύνη του ΦΡΑ. Ε, στη Ρουμανία υπάρχει, έχει αλλάξει πολύ η κοινωνία ε, και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ζήτησε να γίνει ένα δημοψήφισμα ούτως ώστε να μπει στο Σύνταγμα της Ρουμανίας ένας ορισμός της οικογένειας που θα αφασίζεται στη φυσική της μη. Όπως γίνεται και στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, στην Τσεχία, στην Κροατία και στη Σλοβακία. Αυτή η πρωτοβουλία είναι κοινωνικής προέλευσης. Από την κοινωνία την ίδια προέρχεται. Αλλά προσέκρουσε στην αντίδραση και κάποιων ε, τμήματων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ας πούμε. Εμείς δεν θα πρέπει να έχουμε τέτοιες αντιδράσεις. Κάθε λαός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ζητάει να εφαρμοστούν στη χώρα του μηχανισμοί οι οποίοι λειτουργούν καλά αλλού. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα έτσι συμπεριφορών, ας πούμε, ε, αντίθετον προς ε, καλά πρότυπα, ας πούμε. Παραδείγματο χάρη ε, πρωτοβουλίες κατά των διαφόρων νομοθετικών ε, κινήσεων της ε, Πολωνίας. Παραδείγματο χάρη, πριν από λίγα χρόνια ε, υπήρχε μία πρωτοβουλία για να σταματήσουν οι εκτρώσεις. Κάνουμε και τέτοιες συστάσεις μερικές φορές ή ψηφίσματα. Τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτά τα ψηφίσματα. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε, ας πούμε, νομοθετικές πρωτοβουλίες άλλων χωρών. Άλλα παραδείγματα. Υπάρχει ένα ψήφισμα το οποίο αφορά μία νομοθετική πρωτοβουλία από 900.000 πολίτες κατά της, ε, των αυλώσεων. Ακόμα και εκεί υπήρξε αντίδραση εναντίον αυτής της πρωτοβουλίας των ε, πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών θεωρείται ως απειλή στην υποτιθέμενη, ας πούμε, η λεγόμενη δημοκρατία. Σε αυτές τις περιπτώσεις που σας ανέφερα, στην πραγματικότητα τι διακυβεύεται. Το δικαίωμα στη ζωή και το δικαίωμα στην οικογένεια. Βάλουμε εναντίον αυτών των δικαιωμάτων. Και είναι περίεργο με βάση απαντήσεις που μου έδωσε και η Κομισιόν. Δηλαδή, εκεί δεν δράει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί μιλάει, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό είναι ελεύθερη επιλογή και ελεύθερη βούληση των κρατών μελών και των πολιτών. Όμω, όταν υπάρχει μια πρωτοβουλία πολιτών που προτείνει συγκεκριμένε νομοθετικέ δράσει, τι γίνεται, πώ αντιδρούμε εμεί. Θα πρέπει η υπηρεσία σα, ο οργανισμό ΦΡΑ, να γνωρίζει ε, και αυτά τα προβλήματα και να χρησιμοποιεί την έγκλη που έχει, το κύρος που έχει, ούτω ώστε να σταματήσουμε να προσπαθούμε να σταματήσουμε το γεννάστε τέτοιες πρωτοβουλίες. Να φημώσουμε, να προκαλέσουμε ασφυξία σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Ε, και τελικά ακούγονται μόνο τα κόμματα τα οποία έχουν φωνή και στα ΜΜΕ. Τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες, ας πούμε, τέτοιου τύπου άνθρωποι τελικά δεν έχουν φωνή. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον ε, εκπρόσωπο της ΦΡΑ για την πολύ πλατιά και πλήρη παρουσίασή του. Καταρχάς, κάτι που είπε ο κύριος Μπόνι για το LGDPR. για το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Φυσικών Προσώπων και για το κατά πόσον ε, γνωρίζουν τα άτομα ε, τα δικαιώματά τους και κατά πόσον υπάρχει ακρίβεια, πούμε, σε όλο το σύστημα. Ε, χρήσιμες ερωτήσεις ήταν αυτές σχετικές, και, όμως το απορρέον ερώτημα είναι, πιστεύουμε ότι με την εφαρμογή του κανονισμού αυτού μπορούμε να ξεπεράσουμε κάποια από τα προβλήματα. Σε ό,τι αφορά την γνώση των δικαιωμάτων μας, ε, που υποτίθεται θα μας βοηθήσει ο κανονισμός για να τα μάθουμε. Επίσης, για το φόρουμ το για τα, ανθρω... για τα θεμελιώδη δικαιώματα να σας συγχαρώ. Βλέπουμε όλο και περισσότερα κράτη-μέλη όπου, όπως και στη δική μου χώρα ας πούμε, ε, όλοι θεωρούν ότι πρέπει να έχει κανείς, ας πούμε, μία και μόνη ταυτότητα, τη δική, την εθνική του ταυτότητα, όχι άλλες. Ενώ βλέπουμε σε πιο διεθνές πλαίσιο, σε πιο ενοποιημένο πλαίσιο ή παγκοσμιοποιημένο, οι άνθρωποι έχουν περισσότερες ταυτότητες και εθνικότητες. Και εθνικότητες μάλιστα διαφορετικές από τη δική τους έχουν να κάνουν ταυτότητες αυτές με άλλους τύπους, ε, με άλλες πεπιθήσεις, με το σεξουαλικό προσανατολισμό κτλ. Ε, το θέμα είναι ε, πώς το βλέπουμε το θέμα. Θέλω να να σταματήσει αυτή η ιστορία όπου μονίμως αμφισβητούμε ας πούμε την ε, πίστη κάποιων ανθρώπων ε, και τελικά την ε, προσδιορίζουμε αυτή την ιστορία με πολύ κοντόθωρη σκοπιά. Ε, επίσης υπάρχει το info system για τα θεμελιώδη ε, δικαιώματα. μπορούμε να κλικάρουμε ήδη, ε, μπορούμε να ψάξουμε ένα θέμα και αναχώρα από ό,τι κατάλαβα. Το πρόβλημα μέχρι τώρα ήταν ότι δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε πάνω σε μια συγκεκριμένη χώρα. Τώρα έχετε όλα τα δεδομένα και βλέπω ότι έχει αναφορές και σε άλλους φορείς όπως ο ΙΕ. Θα βοηθούσε πάρα πολύ αυτό ε, στη δουλειά που κάνω εγώ ας πούμε για την Ουγγαρία. Και για το μελλοντικό κοινοβούλιο θα βοηθούσε ας πούμε και στο θέμα της ε, Πολωνίας. Ε, είναι μια καλύτερη εκδοχή λέει, του παλιού συστήματος. για το πολιετές πλαίσιο χρηματοδότησης. Κάνατε παρατηρήσεις για, την, για την, τον οργανισμό θεμελιωτών δικαιωμάτων, για τη λειτουργία της και είπατε ότι δεν έχετε αρκετούς πόρους. Αυτό το θέμα θα πρέπει να λυθεί στα πλαίσια της συζήτησης. Πρέπει να κάνουμε όμως αυτή τη συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για να απαντήσουμε στο ερώτημα αν χρηματοδοτούμε καλά ε, την υπηρεσία σας και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όταν φτάσουμε στις τελευταίες φάσεις διαπραγμάτευσης θα πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα, συνάδελφοι. Να ακούσουμε άλλους δύο μιλητές και εν συνεχεία να δώσω το λόγο στο Μάικλ για να απαντήσει, γιατί έχουμε και τις ψηφοφορίες στη 10. Δύο ακόμα ομιλητές και μετά κλείνω τον κατάλογο. Σας παρακαλώ δείξτε κατανόηση δύο μιλητές και μετά ο Μάικλ. Η κυρία Κιέγγε είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ, Κλοντ, και εγώ ευχαριστώ τον Διευθυντή για την παρουσίασή του. Θέλω να θέσω ένα συγκεκριμένο ερώτημα στο Διευθυντή. Καταρχάς να το συγχαρώ γιατί διάβασα την έκθεση για το 2018-2020 ε, και την βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ αντικειμενική. Τα θέματα τα οποία με ενδιαφέρουν που είναι για τη μετανάστευση και το άσυλο, αλλά και τις διακρίσεις και το ρατσισμό, χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση για να τα διαχειριστούμε όλα αυτά. Και κάθε τομέας, κάθε πτυχή αυτού του φαινομένου που κατά περιόδους γίνεται και μαζικής φύσεως όπως το μεταναστευτικό, δεν μπορούμε να το ξεχνάμε από καιρούς καιρών. Περνάω τώρα στο θέμα που νομίζω θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο. Πριν από λίγες μέρες στην Ιταλία, στην Ματσεράτα, ένας ε, κύριος βγήκε στο δρόμο και πυροβόλησε σε έξι άτομα για να σκοτώσουν ε, όσο να τον περισσότερους μαύρους. Ε, δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, γιατί πριν λίγες μέρες ε, έγιναν δηλώσεις από άτομα τα οποία αρχίζουν να μιλάνε για την υπεροχή της λευκής φυλής. Επί χρόνια στο κοινοβούλιο εδώ ε, λέω ότι θα πρέπει να βάλουμε στη μέση διάταξη το θέμα της αφροφοβίας. Ε, υπάρχει καταπολέμηση της, ε, προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την Ισλαμοφοβία ε, την τσιγκανοφοβία κτλ. Θα ήθελα να αναγνωρίσετε επίσημα τις διακρίσεις που υφίστανται, οι, τα άτομα αφρικανικής προέλευσης. Είναι πολύ σοβαρό το, να μην μπορεί κανείς να βγάλει, να βγαίνει στον δρόμο. Φανταστείτε κάποιον ο οποίος, ας πούμε, βγαίνει στον δρόμο και, και, και πυροβολεί, ας πούμε, αφόους. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα η καταπολέμηση της αφροφοβίας κάπου θα πρέπει να αναφερθεί. Δεν μπορούμε να την θεωρούμε μια απλή διάκριση, γιατί έχει ειδικά χαρακτηριστικά, ειδικό μίσος ανάμεσα απέναντι σε ανθρώπους ε, μαύρους, ε, αφρικανικής προέλευσης κτλ. Είναι πολύ σοβαρό, από λευκούς βεβαίως. Είναι ιδιαίτερη μορφή ρατσισμού και θα πρέπει ε, να έχουμε σαφείς στρατηγικές να κάνουμε προσπάθειες ε, με σχέδια δράσης, συστάσεις προς τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι η συνεισφορά της ΦΡΑ θα μπορούσε να είναι σημαντική εδώ, ειδικά στην φάση συλλογής δεδομένων. Και θα μπορούσε να δώσει ειδική όθηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τη πρόξει, ούτως ώστε να αναγνωρίσει αυτή την ειδική μορφή ρατσισμού. Κλείνοντα, θα ήθελα να σα πω ότι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εγώ θέλω να δημιουργεί και ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σισίλ. Ξέρω ότι το θέμα της, ε, των ε, Αφρικανών θα είναι ένα θέμα που θα απασχολεί στον οργανισμό. Συμφωνώ απόλυτα, λέει η κυρία Γκομές, ε, σε αυτό που είπε η συνάδελφος για το θέμα της αφροφοβίας και σε σχέση με αυτό το έγκλημα που έγινε στη Ματσεράτα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο Ιταλικό προφανώς, είναι ουσιαστικό πρόβλημα <clears throat> και μπορεί να επιδεινωθεί. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την έκθεση. Είναι, ήταν λεπτομερής και πιστεύω είμαι απολύτως πεπισμένη ότι ο οργανισμός δεν έχει επαρκείς πόρους. Παρά τα αυτά, Πράγματι κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Κυρίως ευαισθητοποιήθηκα αυτά, από αυτά που είπατε για το θέμα σε σχέση με τη μετανάστευση. Όχι μόνο για αυτά που κάνετε στα hot spot, αλλά εν γέννη για τη μετανάστευση και τις δυσκολίες που βλέπετε ε, στο πεδίο και στις ε, διαδικασίες που αφορούν την ε, τους ετούντες άσυλο. Την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκα το Ιράν με μια αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου και πραγματικά ντράπηκα όταν μιλάμε για το Ιράν και πολύ συχνά μιλάμε για το Ιράν με αρνητικό τρόπο, αλλά με 80 εκατομμύρια πολίτες το Ιράν εδώ και 50 χρόνια φιλοξενεί πάνω από 3 εκατομμύρια ετούντες άσυλο και ε, πρόσφυγες και έχει το μέγεθος της Γερμανίας. Δίνει άδεια, εξασφαλίζει ε, μόρφωση για όλους, όχι μόνο στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες, γιατί οι περισσότεροι πρόσφυγες είναι Αυγανοί. Και προσφέρει η υγειονομική περίθαλψη. Είναι πραγματικά ντροπή για μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που κάνουμε αυτά που είπατε εσείς. Και αυτό το οποίο άκουσα, ε, άκουσα σήμερα το πρωί τον κύριο Όρμπαν να μιλάει κατά της μετανάστευσης. Ε, πραγματικά είναι γελίο. Γελίο θα έλεγα, πέρα από όλα τα άλλα. Και τέλος θα σας, θέλω να σας ρωτήσω συγκεκριμένα εσείς φροντίζετε τα θέματα που διαδραματίζονται εντός της Ένωσης. Αλλά στα κράτη-μέλη αναθέτουν την ευθύνη στο εξωτερικό, κυρίως στο θέμα της ε, μετανάστευσης, συγκεκριμένα στη Λιβύη. Και πληρώνονται χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων την κατάρτιση η οποία στην ουσία, η οποία στην ουσία είναι ε, κράτηση, βασανιστήρια και ένα σωρό άλλα πράγματα που υφίσταται αυτοί που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη. Έχετε ποτέ την ευκαιρία να πάτε να δείτε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάρτιση των εκπαιδευτών που θα καταρτήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Και επιπλέον, συμφωνώ μαζί σας ε, που για το θέμα ότι ζητάτε περιττέρω αρμοδιότητες εξουσίας, το θέμα της αστυνομική και δικαστικής συνεργασίας ε, επί θεμάτων. Και όταν βλέπω, και αυτό δεν αφορά μόνο μια χώρα, αλλά υπάρχει μια χώρα όπου έχει ε, ε, συνέβη κάτι το φοβερό που δεν συμβαίνει συχνά στην Ευρώπη. Η χώρα αυτή είναι η Μάλτα. Δολοφονήθηκε δημοσιογράφος. Και αυτό αφορά το δικαστικό και το αστυνομικό σύστημα, όπου προφανώς κάποια συμμετοχή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα ήταν ε, πολύτιμη. Θα ήθελα να σας ζητήσω να το μελετήσετε. Υπάρχουν και άλλες ζητήματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του είδους την προσφορά είναι ζητούμενη. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ας ε, πάμε στο Μάικλ τώρα να, κάνει κάποιες, να δώσει κάποιες απαντήσεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή για τις πολύ σωστές ε, ε, ε, ερωτήσεις. Κύριε Κινίτσι, ρωτήσατε πολλές, κάνατε πολλές ερωτήσεις. Όσον αφορά τα παιδιά και το διαδίκτυο και συνολικά το πώς αστυνομεύουμε το θέμα της, του σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. Με τα χαράς μπορώ να σας αναφέρω ότι ο οργανισμός ξεκινά φέτος ένα νέο έργο, φέτος ένα νέο έργο που αφορά αλγοριθμούς, δηλαδή πριν αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα το νέο αυτό πεδίο δράσης, πρέπει να να γνωρίσουμε την τεχνική σκοπιά των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε ε, αλγορίθμους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τεχνολογία blockchain και μια σειρά από άλλα πράγματα. Ολοκληρώνουμε και ένα έργο για την, ε, ε, τον αλφαβητισμό των μέσων ενημέρωσης και την ευαισθητοποίηση παιδιών και ενηλίκων ώστε να ερμηνεύουν καλύτερα αυτά τα οποία βλέπουν στο διαδίκτυο. Τώρα, όσον αφορά την ε, φροντίδα των ε, ανηλίκων στο πλαίσιο του Eurodac, με τα χαράς ε, θέλω να σας πω ότι γνωμοδότησε ο οργανισμός μας συγκεκριμένα επί του θέματος στο Κοινοβούλιο στις 22 Δεκεμβρίου του 2016. Η γνωμοδότηση ήρθε συστηματικά το σύνολο της πρότασης από άποψη συμμόρφωση με ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως το θέμα των παιδιών, περιλαμβανομένου και του θέματος της απαγόρευσης της χρήσης βίας για τη δακτυλοσκόπηση ενό ενός παιδιού, όπως επίσης και τα θέματα της προστασίας. Όσον αφορά την ε, την τρομοκρατία των χωρών και το αυξημένο επίπεδο ε, απέναντι στους μουσουλμάνους και εδώ συνδυάζομαι όσα είπε η κυρία Κιάνγκα για θέμα, ε, ανθρώπους αφρικανικής ε, προελεύσεως καταγωγής. Θέλω να πω ότι αναπτύσσουμε κάτι που φέτος θα ξεκινήσει για να εξασφαλίσουμε ότι το προφίλ το που φτιάχνει η αστυνομία για τα άτομα συνάδει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την ψηφιακή εποχή που το προφίλ πλέον δεν το κάνει ο αστυνομικό, αλλά ένα μηχάνημα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πάρουμε υπόψη μα. Ε, όσον αφορά τον κύριο Μπόνι. Κύριε Μπόνι, ε, ξεκινήσαμε μια έκθεση μια νέα έρευνα μάλλον για τον αντισημιτισμό. Θα γίνει φέτος και θα, θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα το Δεκέμβριο του 2018 και αυτό θα σας βοηθήσει καθώς ε, παρακολουθείτε τις διάφορες μορφές ε, αυξανόμενων της εντός της Ένωσης. Ο κύριος Μπόνι επίσης ρώτησε αν λαμβάνουμε υπόψη μας τις επιπτώσεις επί των πολιτών των αρνητικών κινήσεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι μια από τις βασικές προσπάθειες. Το το, ε, το ε, σύστημα που παρακολουθεί τα θεμελιώδη δικαιώματα θα μας βοηθήσει να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς λέγεται σε αυτό το, σε αυτού του θέματος. Επιπλέον, είναι πρόσδεκτη η πρόταση του κύριου Μπόνι να το Κοινοβούλιο να ε, επανεξετάσει τις συστάσεις μας για την κοινωνία των πολιτών και ε, τακτικά. Θα θέλαμε να, να γίνει αυτή η προσπάθεια. Θα θέλαμε επίσης να σας πούμε ότι κινείται και η Κομισιόν ακριβώς το ίδιο στην διακατεύθυνση ε, σε θέματα χρηματοδότησης. Κύριε Γιούρεκ, ευχαριστώ για τις προτάσεις σας. Υπάρχουν θέματα οικογένειας και αναπαραγωγής όπως η άμβλωση που δεν είναι ε, αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα δεν μπορεί να τα μελετήσει οργανισμός. Κυρία Σαντίνη, όσον αφορά τα ε, σφάλματα που γίνονται με τα βιομετρικά στοιχεία. Στην έκθεση του Απριλίου θα δούμε την μέχρι τούδε πρακτική. Και δεν είναι θέμα ότι φταίει ο κανονισμός ή ο νόμος, είναι φταίει η εφαρμογή. Και βεβαίως η, κακή εφαρμογή θα ε, εξακολουθήσει να ισχύει και μετά τη θέση ενισχύει της οδηγίας GDPR. Επίσης, ε, θέλουμε να δημοσιεύσουμε ένα εγχειρίδιο για αυτούς που ζητούν προστασία δεδομένων. Το, θα το ε, εκδώσουμε τον Μάιο που θα τεθεί ενισχύει η οδηγία. Επίσης, το θέμα του ε, ε, ανίκην είναι ακριβώς, ε, έχει ακριβώς την ίδια έννοια με αυτή που παρουσιάσατε εσείς. Τώρα, όσον αφορά την έλλειψη πόρων, πράγματι ε, θα επιστρέψουμε στα μέλη του Κοινοβουλίου με συγκεκριμένες αναλύσεις και προτάσεις για το πώς μπορούν να προστατευθούν καλύτερα τα θεμελιώδη δικαιώματα μέσω του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου. Κυρία Κιάνγκε, με χαρά σας ε, ενημερώνω ότι στις 28 Νοεμβρίου θα δημοσιευθεί μια έκθεση με βάση την έρευνα EU Midas που έχει τίτλο «Μαύρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και θα αναφέρει την εμπειρία ε, ανθρώπων από την υποσαχάρια Αφρική και τις εμπειρίες του και θα αναφερθεί ακριβώς σε αυτά τα θέματα που θέσατε. Κυρία Γκόμες, τέλος περιορίζουμε, έχουμε περιορισμένη δυνατότητα να κοιτάξουμε εκτός της γεωγραφικής επικράτησης Ένωσης. Μπορούμε να το κάνουμε. Το κάναμε στην έκθεση για τα βιομετρικά στοιχεία. Θέλουμε να δούμε τι γίνεται στις πρεσβείες Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της χώρας. Εκεί συγκεντρώνουν τα δεδομένα για να μπουν στα αυτά τα, τα μεγάλα συστήματα. Η, το, το Κοινοβούλιο ε, που ε, ε, αναπτύσσει έναν κατάλογο ασφαλών χωρών επιστροφής. Αλλά το θέμα αυτό για τις χώρες που αναφέρατε εσείς είναι εκτός των δυνατοτήτων μας. Και ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις όσον αφορά τη Μάλτα. Σαφώς θα μελετήσουμε το θέμα περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Μάικ. Ευχαριστώ και για τη συντομία γιατί βλέπεις ότι έχουμε ψηφοφορίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα πω τα τετριμένα. Ε, τονίζουμε και πάλι τη σημασία των διαπροσωπικών επαφών των βουλευτών με τον οργανισμό και επίσης αυτό που είπε ο κύριος Μπόνη, ε, τι συνέχεια δίνουμε στις ε, εκθέσεις σας και επίσης και τους δείκτες που μπορεί να χρειάζεται στο μέλλον κτλ. Εντάξει, ε, συνεχίζεται πάντως η υπόθεση αυτή, δεν σταματάει εδώ, θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε για την εξαιρετική έκθεση και την εξαιρετική δουλειά που κάνεις εσύ και οι ε, συνεργάτες. Λοιπόν, αν είστε έτοιμοι να ψηφίσουμε συνάδελφοι, καθίστε σας παρακαλώ. We, um, So we have the opinion on the annual report. Λοιπόν, έχουμε την ετήσια έκθεση του 2016 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά πολέμηση της απάτης. Η κυρία ε, Κουντρίτσκα είναι η συγκεκριά. Μπάρμπαρα, θέλεις να λάβεις το λόγο για ένα λεπτό. Έχουμε ε, πολλές συμβαστικές ε, τροπολογίες και σας συνιστώ να υπερψηφίσετε παρακαλώ τις τροπολογίες αυτές. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους ε, ε, τους και οδησηγητές, τη γραμματεία και τους συμβούλους μας. Ωραία. Ψηφίστε την έκθεσή μου και ευχαριστώ. Κατάλαβα το μήνυμα. Ελήφθη over. Τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάρβαρα. Είστε έτοιμοι. Συμβαστική ένα Αρχίζει η ψηφοφορία τώρα. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. στην ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 9. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 10 και 11 ταυτίζονται, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 12, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Συμβαστική 3, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 16 αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 22 αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. 4 διορθώνει ο πρόεδρος, συγγνώμη. Συμβαστική 4 ψηφίζουμε. Ευχαριστώ, Τόμας Στεχόφσκι. Ε, εγκρίνεται. Η συμβαστική 5, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 27, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρα. Επίση εγκρίνεται και τώρα η τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα παρακαλώ. Εγκρίνεται 39 ψηφί υπέρ, 8 κατά και 3 αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Κούντριτσκα. Ολοκληρώνονται οι ψηφοφορίες συνάδελφοι εδώ. Ο κύριος Ράντεφ. Um, Συνάδελφοι, έλεγα να συνεχίσουμε και παρακαλώ αποχωρήστε ησύχως αν μπορείτε. Επόμενο θέμα είναι δύο θέματα. Όχι, παραπάνω μέχρι 14 κοινή συζήτηση για τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Barbados για την τροποποίηση συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ε, και των Barbados σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης ε, για βραχία διαμονή και ακολουθούν και άλλες χώρες, ε, ο Μαυρίκαιος κλπ. Θα τα δούμε αυτά. Το λόγο έχει ο κύριος Πάβελ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ω εισηγητής σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου για ε, συμφωνία με ε, έξι ε, χώρες εταίρους, οποίες δεν πρόκειται να σας αναφέρω, τις ξέρετε. Πρώτα αξιολογείται η κατάσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνίες με τις έξι αυτές χώρες για ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς θεώρηση διαβατηρίου των πολιτών της Ένωσης και των υπολείπων Ε, για 90 μέρες ε, εντός ενός εξαμήνου αλλάζει αυτό την προηγούμενη συμφωνία ε, και με τις Μπαχάμες για τη βίζα βραχιάς διαμονής. Επίσης, η δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει γίνει πλέον Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2009 από την συνθήκη της Λισαβόνας και η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον έχει νομική προσωπικότητα. Επίσης θα ήθελα να σημειώσω ότι η άρση υποχρέως θεώρησης ε, αφορά ε, όλους ε, τους πολίτες και διπλωμάτες και κατόχους ειδικών διαβατηρίων για όλες τις κατηγορίες και όλες τις δραστηριότητες με μια εξαίρεση για εμβάθυνση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εξευθέ χώρες. Έχουμε πολιτικό διάλογο με χώρες ΑΚΕ και ιδιαίτερα αυτές τις χώρες που είναι χώρες ΑΚΕ που εντείνεται και αυξάνεται. Αυτή η συμφωνία για την άρση θεωρήσεων ε, εγγράφεται στο πλαίσιο της συνέχισης ε, των σχέσεών μας και θα εκπέμψει ένα θετικό μήνυμα υποστήριξης προς τις χώρες αυτές και τις προσπάθειες που κάνουν. Θέλω επίσης να επιστήσω την προσοχή σα. Ε, στη μεγάλη συμμετοχή της ε, Κροατίας, ε, Κύπρου, Ρουμανίας και Βουλγαρίας για την ε, ολοκλήρωση του χώρου Σέγγεν. Έχω πει και στην έκθεσή μου ότι αυτό θα πρέπει το σύντομότερο να έχουν διμερείς συμφωνίες συνάψει όλες οι χώρες και ως προς το χρονοδιάγραμμα 26 Φεβρουαρίου η προθεσμία κατάσταση τροπολογιών. Συνεδριάσεις θα γίνουν μόνο εφόσον απαιτούνται. Να δούμε και τις τροπολογίες στην Επιτροπή. Θα δούμε πότε θα ψηφίσουμε. Θα μας τα πείτε εσείς Πρόεδρε αυτά. Και θα εγκριθεί μάλλον στην Ολομέλεια το Μάιο ή τον Ιούνιο. Thank you very much, And just Ευχαριστώ πολύ. Ε, είστε εισηγητής για τις έξι χώρες αυτές και συστάσεις. Είναι διαδικασία ε, σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω, θέλει κανένας από τους κοιόδης να πάρει το λόγο. Η κυρία Βαλέρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, δεν θα μακρηγορήσω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και μια αντίρρηση για τις εκθέσεις αυτές. Είναι όλο και περισσότερες οι χώρες που ε, χαίρουν αυτού του καθεστώτος. Μια παρατήρηση μόνο θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Η άρση θεωρήσεων σημαίνει, υποχρέωση θεώρησης δηλαδή, σημαίνει για κάποιες χώρες ότι θα πρέπει να ε, χρησιμοποιήσουν ένα συγκεκριμένο σύστημα ε, Και γιατί το αλλάξαμε το σύστημα, μήπως αυτό είναι κρυφή ε, επαναφορά της θεώρησης διαβατηρίων. Ευχαριστώ. Ο Ισκιώδης ε, των Πρασίνων και του Άλτε, κυρία Λούντε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Κύριε Πάβελ, συγχαρητήρια που δουλέψατε σε αυτό το ε, θέμα της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Όσον αφορά την απελευθέρωση των θεωρήσεων για τις χώρες που αναφέρατε, θέλω να πω ότι η απαλλαγή ε, από την υποχρέωση θεώρησης για βραχία διαμονή είναι σημαντικό εργαλείο. Οφελεί τους πολίτες, ενθαρρύνει την, τον διαπολιτισμικό διάλογο, την κατανόηση και το αίσθημα του ανήκει σε έναν κόσμο χωρίς σύνορα. Θα ήθελα όμως να κάνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας κατά νου πόσο σημαντικό είναι το Κοινοβούλιο ως συνομοθέτης. Να ζητήσω περισσότερη διαφάνεια στην ε, προετοιμασία των συμφωνιών αυτών των ε, απαλλαγών θεωρήσεων για βραχίες διαμονές. Θα έπρεπε να είχα, μας είχαν δοθεί περισσότερες πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία, μεγαλύτερες διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ολόκληρη τη φάση, αλλά κυρίως πριν συναυθούν αυτές οι συμφωνίες και όχι εκ των υστέρων. Ευχαριστώ για το έλκο, κύριος Ράντεφ. Ευχαριστώ για το λόγο κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι συμφωνίες για την ε, απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση για βραχία διαμονή για τους πολίτε των χωρών αυτών δείχνει πόσο έχει δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην οικονομική και πολιτική ανάπτυξη των χωρών οι συμφωνίες απλώς πρέπει να ενημερωθούν με βάση τις εξελίξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Συμφωνώ με τη σύσταση του κυρίου Πάβελ φυσικά να πούμε ναι, να συνενέσουμε στις συμφωνίες αυτές. Παρά τα αυτά θέλω να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει τις συμφωνίες εγκαίρως. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνενέσει πριν τεθούν ενισχύει οι συμφωνίες και όχι ένα χρόνο αργότερα. Αυτό θα ήταν μια πολύ συναδελφική στάση μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων και ελπίζω ότι αυτό το πνεύμα θα επικρατήσει στο μέλλον. Κάτι άλλο που θέλω να θέσω. Οι συμφωνίες πρέπει και πάλι να τροποποιηθούν ώστε να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία θα ενταχθούν στο σύστημα εισόδου-εξόδου. Αυτό συμφωνήθηκε πέρσι και θα αρχίσει το σύστημα να λειτουργεί το 2020. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται από αυτό. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει άλλος σκιώδης αν δεν κάνω λάθος, οπότε ο κύριος Παύλ και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Α, η κυρία Βεργιέ. Δεν με βλέπετε κύριε Πρόεδρε και παρόλα αυτά είμαι κατευθείαν απέναντί σας. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Ε, βρίσκομαι εδώ από το 2009, άρα έχω μια συνολικότερη προσέγγιση. Η ομάδα μου εκφύσεως είναι υπέρ της απελευθέρωσης των θεωρήσεων για τους λόγους που ανέφερε ο συνάδελφος από την ομάδα των φιλελευθέρων. Θα ήθελα να επιμείνω στο ότι η πολιτική αυτή είναι μια μεταβλητή γεωμετρία. Οι χώρες αυτές ε, είναι πολύ ενδεικτικές. Είναι χώρες επί για τις οποίες η απελευθέρωση των θεωρήσεων θα διευκολύνει περισσότερο τους Ευρωπαίους ε, γιατί πρόκειται για εξαιρετικούς προορισμούς διακοπών, άρα η απελευθέρωση θεωρήσεων θα χρησιμοποιηθεί ε, όχι για σκοπούς πραγματικά εταιρικής σχέσης δεν θα σας εκπλήξει, κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ στους ε, τινήσιους, οι οποίοι έχουν τεράστιες δυσκολίες να ξεκινήσουν πραγματεύσεις εποφελία και των δύο εταίρων. Συμφωνώ με αυτό που αναφέρθηκε στο θέμα της διαφάνειας και την ανάγκη, για την ανάγκη να γίνονται σεβαστές οι ευρωπαϊκές συνθήκες. Δηλαδή το Κοινοβούλιο να εμπλέκεται εκ των, εκ των, εκ των προτέρων. Η κυρία Γκαμπριέλ που από καιρό ήταν ε, εισηγήτρια από αυτού, επενελειμμένος έχει υπογραμμίσει το στοιχείο και πιστεύω ότι θα συνεχίσει, πρέπει να συνεχίσει να ε, επιμένει. Δάλλως ε, γελιοποιούμε το Κοινοβούλιο και τα δικαιώματά του αν ερχόμαστε εκ των υστέρων να ενημερωθούμε. Πρέπει εκ των προτέρων να ενημερωνόμαστε για την... πριν δηλαδή τεθούν ενισχύ συμφωνίες. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Thank you, Marie Ευχαριστώ Μαρή Κριστίν. Ε, Εμίλιαν, ήθελε να πάρει το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω όλου του χιώδη ομιλητέ για τα σχόλιά του και προσβλέπω στην ψηφοφορία. Άννα, ήθελες το λόγο. Σύντομα παρακαλώ. Θέλω απλώς να συμφωνήσω, να στηρίξω με αυτά που είπε η Μαρή Κριστίν Βερζιά στην προειδοποίηση που διατύπωσε ότι πρέπει να βλέπουμε μόνο έτσι τα θέματα. Οι χώρες αυτές είναι χώρες που είναι πολύ σημαντικές ε, στο ξέπλυμα χρήματος. Και όχι μόνον. Ας πούμε ο Άγιος Χριστόφορος και Νέβης εμπλέκεται σε ένα μεγάλο σκάνδαλο με εταίρους που εμπλέκονται σε κάποιες από τις ευρωπαϊκές χώρες μας, περιλαμβανομένης της δικής μου και κυρίως στη Μάλτα, εμπλέκονται σε αυτό το πρόγραμμα πωλήσεως ευρωπαϊκής Ιθαγένειας και ευρωπαϊκών διαβατηρίων για σκοπούς ε, ξεπλήματος χρήματος. Ο Άγιος Χριστόφορος και Νέβης είναι μια χώρα όπου υπάρχει η ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα εμπλέκεται σε ένα τεράστιο πρόβλημα επειδή χρησιμοποιείται το σύστημα για μεγάλο, μεγάλα προγράμματα ξεπλήματος χρήματος ανθρώπων οι οποίοι θεωρούν ότι είναι ε, ε, πολίτες του κόσμου, δηλαδή εύποροι οι οποίοι πηγαίνουν εκεί με πλούτο που έχει αποκτηθεί καλά ή λιγότερο καλά από διάφορα μέρη του κόσμου από φορολογικές, ε, για να φύγουν από φορολογικές αρχές και για να κρύψουν κατά καιρού ε, έσοδα από εγκληματική δραστηριότητα. Άρα θα ήθελα να είμαστε προσεκτικοί, επιφυλακτικοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση και φυσικά τον εισηγητή η προθεσμία ε, τροπολογιών 26 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Και τώρα έχουμε μια δυσκολία, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί είμαστε λίγο νωρίς. Έχουμε... Το επόμενο θέμα ε, προγραμματίζεται για τις 11 παρα 20 κανονικά, που αφορά την ε, αναδιατύπωση των ηλεκτρονικών συστημάτων διοδίων. Είναι όλοι εδώ όσοι εμπλέκονται με το θέμα. Ο εισηγητής της γνωμοδότησης είναι εδώ, κύριος Σκρίπεκ. Θα διακόψουμε λοιπόν μέχρι τις 11 παρα 20. Επειδή ο εισηγητής δεν έχει έρθει ακόμα, σας παρακαλώ να διακόψουμε μέχρι τις 11 παρα 20. Να επιστρέψετε γέρος, αν θέλετε να συμμετέχετε στη συζήτηση του 16 για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων. Ευχαριστώ. Διακόπτουμε μέχρι τις 11 παρά 20. Ευχαριστώ. Περιμένουμε για να κάνουμε το θέμα για τη διαλειτουργικότητα. Τελικά θα αρχίσουμε στις 11 η ώρα. Ζητώ συγγνώμη που θα καθυστερήσουμε περαιτέρω. Ζητώ συγγνώμη ε, απέναντι στους βουλευτές και στους α, υπαλλήλους. Στις 11 θα με αντικαταστήσει ο συνάδελφος θα ξεκινήσουμε στις 11 με το σημείο 16 για τη διαλειτουργικότητα. Ευχαριστώ, θα το πω και στους συναδέλφους που είναι έξω, ότι θα ξεκινήσουμε στις 11. ιδιαίτερα Υπότιτλοι Με κάποια μικρή καθυστέρηση, συναδελφοί, θα ξαναρχίσουμε την, ε, τη συζήτησή μας. Το επόμενο σημείο είναι η διαλειτουργικότητα των συστημάτων ε, τηλεδιοδίων και η διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής κτλ. κτλ. Της 31 Μαΐου του 2017 η Κομισιόν δημοσίευσε την ε, πρόταση οδηγίας που αφορά μια αναδιατύπωση και η Επιτροπή Τραν είναι η καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή και στις 22 ε, Ιουνίου οι συντονιστές της ΛΥΜΠΕ αποφάσισαν να εκδώσουν μια γνωμοδότηση. Ο εισηγητής είναι ο κύριος ε, Σκρίπεκ. Υπάρχουν ε, ερωτήσεις. Ε, πάντως η Γενική Διεύθυνση ΜΟΥΒ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παρούσα και θα μπορούσε να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις σε περίπτωση που έχετε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σκρίπεκ για να παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την ε, Κομισιόν για την πρότασή της που υποβλήθηκε κατά την παρουσίαση της ε, αναδιατύπωσης της οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδίοδιων. Είναι ξεκάθαρο ότι η ελεύθερη κυκλοφορία έχει φέρει νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις, ειδικά στον τομέα των μεταφορών, ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία από τις προθέσεις της αναδιατύπωσης της οδηγίας είναι να ανοίξει η αγορά για ηλεκτρονικά διόδια, ούτω ώστε να μπορούν να λειτουργούν σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υπάρχει με ένα μηχάνημα ε, σε κάθε όχημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε ε, να διευκολυνθεί όλο το σύστημα και να λειτουργεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, θα ήταν πρακτικό για τους επιχειρηματίες και για τους πολίτες. Η πρόθεση είναι να υπάρχει ένα σύστημα με μία ηλεκτρονική συσκευή που θα δίνει δυνατότητα στον οδηγό να ταξιδεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να σταματά στα διόδια. Και τα διόδια τα πληρώνει ηλεκτρονικά, απευθείας. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ απλό. Ο απλός πολίτης λοιπόν ε, θα μπορούσε να τα πληρώσει έτσι. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, αλλά θα διευκόλυνε πάρα πολύ τα πράγματα. Προς το παρόν υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα εφαρμοστεί κάτι τέτοιο όμως, ούτω ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω η ενιαία αγορά. Στην κνομοδότησή μου εστιάζω κυρίως στο στην περίπτωση που δεν γίνεται καταβολή των ηλεκτρονικών διοδίων, α, των τηλεδιοδίων, αυτό είναι πρόβλημα το να μην καταβάλει κανείς τα διόδια, γιατί θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε ε, τότε το σύστημα μεταξύ των κρατών μελών ε, λόγω μη συνεργασίας. Η αναδιατύπωση προτείνει ότι σε περίπτωση μη πληρωμή σε κάποιο κράτος μέλος, οι πληροφορίε ε, και τα δεδομένα θα κυκλοφορήσουν, ούτω ώστε να εντοπίσουμε την ταυτότητα του κατόχου του οχήματος. Στην ε, τροπολογία μου προτείνω ότι είναι σημαντικό να διακρίνουμε ανάμεσα σε μια χώρα όπου η μη καταβολή των ε, τηλεδιοδίων είναι ποινικό αδίκημα. Σε αυτή την περίπτωση διευκολύνονται οι ποινικέ διαδικασίες, αλλά σε χώρες όπου το αδίκημα αυτό είναι απλώς διοικητικό παράπτωμα, ε, σαν να πληρώνει κανεί, να πληρώνει το, την κλίση του, α πούμε, για παράνομο παρκάρισμα, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πληρωθεί ένα απλό πρόστιμο. Θα πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στα δύο συστήματα, δηλαδή ποινικό αδίκημα ή διοικητικό. Οι χώρε οι οποίε υφίστανται ζημία γιατί δεν μπορούν να, ε, να επιβάλλουν την ε, πληρωμή, το χάρη στη Σλοβακία, Εάν ε, χάρη στην αναδιατύπωση της Κομισιόν ε, υποχρεούνταν όλοι να πληρώνουν, ε, θα καλύπτονταν τα κενά. Θα πρέπει να γίνουν λοιπόν σε κά, κάποιες αλλαγές στο κείμενο της Κομισιόν και στη δική μου πρόταση προτείνω ε, να ληφθούν μέτρα με απόλυτη συμμόρφωση και σεβασμό του Γενικού Καονισμού για τα προσωπικά δεδομένα θα ανταλλάσσονται προσωπικά δεδομένα και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο μέσα σε, μια συγκεκριμένη προθεσμία για συγκεκριμένο σκοπό. Δηλαδή για να εξασφαλίσουμε την καταβολή των τηλεδιοδίων. Αυτό αφορά ήδη, ισχύει ήδη ε, και για οδηγούς που οδηγούν επικίνδυνα Παραδείγματο χάρη οδηγού οι οποίοι οδηγούν με, υπό την επίρρεια αλκοόλ και τα λοιπά. Θα πρέπει να ισχύσει λοιπόν και για τα ηλεκτρονικά θέματα και για την, τα τηλεδιόδια. Θα πρέπει χάρη στην σωστή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών, να εξασφαλίσουμε την καταβολή των τηλεδιοδίων. Πιστεύουμε ότι την ευθύνη θα πρέπει να την κρατήσουμε στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο λόγω αναλογικότητας και επικουρικότητας, χωρίς υπερβολικό άχθος, χωρίς υπερβολικό διοικητικό άχθος, νομίζουμε ότι μπορούμε να έχουμε τελικά ένα πολύ πιο αποτελεσματικό σύστημα. Εάν διευρύνουμε το σύστημα για να συμπεριλάβουμε και τα πρόστιμα για το παρκάρισμα θα ήταν ακόμα καλύτερα. Αν όμως σε ένα κράτος μέλος η μη πληρωμή των διοδίων θεωρείται ποινικό αδίκημα, τότε θα πρέπει το θέμα αυτό να αντιμετωπιστεί στο επίπεδο εκείνου του κράτους μέλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως ε, τον Γιώσεφ Νάτσο, ο οποίος ε, υπέβαλε πολύ χρήσιμα σχόλια. Και είμαι πεπισμένο ότι οι τροπολογίες των συναδέλφων θα εμπλουτίσουν την πρόταση και αν τα εφαρμόσουμε όλα αυτά, εάν το σύστημα γίνει πιο αποτελεσματικό, τότε νομίζω ότι θα ήταν επωφελές και για τα κράτη-μέλη και την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξεχνάμε ότι η ενιαία αγορά μας δίνει και αυτή τη δυνατότητα. Και λογικό είναι να, πληρω... να τιμωρούμε εκείνους που δεν σέβονται τους κανόνες. Υπάρχουν δύο σκιώδεις συζητητέ μέσα στην αίθουσα. Ε, δεν ξέρω αν άλλοι συνάδελφοι πέρα από αυτούς θέλουν να θέσουν ερωτήματα, να κάνουν κάποιο σχόλιο. Όχι, από ό,τι βλέπω. Παρακαλώ. Λέω κύριο Σούγκουρ. Ε, χαίρομαι για την πρωτοβουλία της Κομισιόν για να αντιμετωπιστούν τα κενά του συστήματος για να γίνει πιο αποτελεσματική η σημερινή νομοθεσία. Δεν νομίζω ότι υλοποιεί τους περισσότερους από τους στόχους της. Σε ό,τι αφορά τις ε, αρμοδιότητές μας σε σχέση με την αναδιοτύπωση της οδηγία και την ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων και το δικαίωμα στην ιδιωτική σφαίρα. Χαίρομαι που υπάρχει ειδική έμφαση από τον ε, εισηγητή στο άρθρο 16 τη συνθήκη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σημαντικό τα, να σέβονται την προσωρινή φύλαξη των δεδομένων, ε, τη χρήση ε, τους επίσης με βάση ε, την αρχή της αναλογικότητας και επικορικότητας. Χρήσιμο θα ήταν να αφαιρθεί και η δυνατότητα να έχουμε εθνικά σημεία επαφής, ούτω ώστε να δίνουν, ε, δίνουν πληροφορίε σε περίπτωση σημείο καταβολή των τηλεοδίων. με βάση τον ορισμό του 2β, ε, θα μπορούσαν επίσης ε, οι εταιρείες τηλεοδιοθήτων να είναι και ιδιωτικές εταιρείες. Και έχει το δικαίωμα να πάρει τις απαραίτητες πληροφορίες ως ιδιωτική εταιρεία για την ε, ανάκτηση των μη καταβληθέντων. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε περαιτέρω συζητήσεις με τον εισηγητή ε, γιατί θέλει να περιορίσει τις δυνατότητες της ε, Κομισιόν να υιοθετεί ε, καταξιόδηση πράξης μόνο σε πέντε χρόνια. Οι μηχανισμοί για την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών ε, βασίζεται γενικά σε, μια διάταξη της οδηγίας του 2015-2013 για την διασυνοριακή εφαρμογή των αδικημάτων που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια. Με βάση αυτήν την οδηγία, η Κομισιόν έχει δυνατότητα να υιοθετεί κατεξουδότηση πράξη για πέντε χρόνια. Όμως, αυτή η οδηγία αναφέρει ότι η εκχώρηση των εξουσιών ε, επεκτείνεται για περιόδους ίδιας διάρκειας, εάν το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν έχουν αντίρρηση. Ευχαριστώ. Κυρία Μαρία Γκραπίνη τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Μπριγκίτα. Είναι πάρα πολύ σημαντική η έκθεση αυτή. Είμαι ικανοποιημένη που η Κομισιόν έχει εγγύψει επί του θέματος. Συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την επικουρικότητα και την αναλογικότητα σε όλες τις εκθέσεις. Επίσης όμως θα πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μόνο οι χρήστες πληρώνουν αυτά τα διόδια. Έχω μια ερώτηση ως προς αυτό. Θα ήθελα να εκφράσω τη θέση και της ομάδας που εκπροσωπώ επίσης. Εάν τα πρόστιμα και οι κυρώσεις διαφέρουν από κράτος σε κράτος, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους ε, επιχειρηματίες να γνωρίζουν αυτές τις διαφορές. Ένας, μια μικρή εταιρεία, πούμε. πώς ξέρει τι συμβαίνει στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να εντυπωσιαστεί και από τις διαφορές ε, στις κυρώσεις. Παραδείγματος τα πρόστιμα ε, επιβάλλονται σε μια χώρα, ενώ σε μια άλλη χώρα μπορεί να επιβάλλεται ποινή φυλάκισης. Υπάρχουν εμπόδια για τις ε, εταιρείε. Δεν μπορούν να ξέρουν τους διαφορετικούς κανόνες σε όλα τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η αλλαγή θα υλοποιήσει το σκοπό για τον οποίο ε, υποβάλλεται. Θα φέρει μεγαλύτερη σαφήνεια και ομοιογένεια. Δεν θα δημιουργήσει μεγαλύτερο κόστος όμως. Συζήτησα με, τις, ε, με ε, διαφόρων εταιριών για το θέμα αυτό και δεν έχουμε βρει καλά μέτρα για να αποφύγουμε την μη κατεβολή των τελών. Πώς θα είμαστε σίγουροι ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Μετά από διαβουλεύσει με συναδέλφου ε, της ομάδας μου, θα υποβάλω τροπολογίες μέχρι τι 26 και ελπίζω να βρούμε ένα καλό συμβασμό ούτως ώστε να βελτιώσουμε την πρόταση της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σίπελ. Δεν έχω δει άλλο συνάδελφο να ρωτάει, να θέλει να ρωτήσει. Παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει σε κάποιες από τις ερωτήσεις της κυρίας Γκραπίνη και αν θέλει να ξαναμιλήσει ο εισηγητής μας. Το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριο Σιουσίκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Δύο πράγματα, αν μου επιτρέπετε, ήθελα να πω για την έκθεση. Νομίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ουσιαστικότατη. Γι' αυτό καλωσορίζουμε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, και δύο σημεία να αναφέρω όπου διαφωνώ με τη γνωμοδότηση. Το πρώτο έχει να κάνει με την πρόταση να υπάρξει διπλή νομική βάση. Αυτό κανονικά είναι εξαίρεση στον κανόνα. Και ακούω ότι η εστίαση στο συγκεκριμένο θέμα είναι ε, στις μεταφορές. Οπότε για ποιο λόγο να χρειάζεται νομική βάση διπλή. Και δεύτερον, το, η παράγραφος 4 στην γνωμοδότηση αναφέρεται ε, στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να πλαισιώνεται και από την νομοθεσία όχι μόνο ε, αυτή καθ' αυτή για τα τηλεδιώδη αλλά και καλύτερη εφαρμογή της. Ε, έρχομαι στην κυρία Γραπίνη. Αυτό που λέτε δεν ισχύει μόνο για τα διόδια, όπου οι εταιρείε ή οι πολίτες άλλων κρατών δεν γνωρίζουν ποια είναι τα πρόστιμα. Αν πας να χτυπήσεις κάποιον σε μια χώρα μέλος, δεν ξέρεις απαραίτητο ποιο είναι το πρόστιμο ή η κύρωση. Δεν πρόκειται μόνο για τα διόδια δηλαδή. Το θέμα είναι να βλέπουμε ποιος είναι ο δράστης ή ο παραβάτης και δεν νομίζω ότι με βάση την επικουρικότητα και τη σχετική αρχή έχουμε το δικαίωμα εμείς να προτείνουμε πλήρη εναρμόνιση των προστίνων. Υπάρχει ένας γενικός κανόνας να είναι ανάλογα ε, με την παράβαση και τα πρόστιμα. Αυτό ισχύει για όλα. Και είναι και φυσιολογικό. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να στραφούμε προς την πλήρη εναρμόνιση των τιμών παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank you. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, Πρόεδρος. Κύριε Σκρίπεκ, θέλετε να επανέλθετε, όχι, έτσι, ωραία. Καλώς. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για την προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών 26 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Θυμηθείτε παρακαλώ ότι πρόκειται για πρόταση αναδιατύπωσης σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού μας. Είναι υποχρεωτικό να δικαιολογείτε τις τροπολογίες σας, αν κάνετε τροπολογίες στο κωδικοποιημένο, το λευκό τμήμα της πρότασης. Μόνο εκείνες οι τροπολογίες ε, που είναι απαραίτητες και έχουν να κάνουν με την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέονται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες θα γίνουν δεκτές. Μόνο αυτές τροπολογίες. Και για να μεταφραστούν οι αιτιολογήσεις δεν θα πρέπει να υποβαίνουν τους 500 χαρακτήρες. Ωραία. Τελειώσαμε με την πρωινή αυτή συνεδρίαση. Δεν ξέρω αν θέλει ο Γιώζεφ Βάιντεν να πάρει το λόγο. Όχι το λόγο, να προεδρεύσει. Έλα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Προχωράμε λοιπόν με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατάσταση του συστήματος πληροφοριών Schengen. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κοέλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, στις 6 Νοεμβρίου η Επιτροπή ενέκρινε τη θέση του Κοινοβουλίου για την αναμόρφωση του συστήματος πληροφοριών Σέγγεν. Θα επικεντρωθώ σε δύο μόνο από τους τρεις φακέλους. Τις εντολές και την αστυνομική συνεργασία. Η πρώτη πήγε κατευθείαν στον τριμερή διάλογο επί Εσθονικής Προεδρίας στις 16 Νοεμβρίου με την ευκαιρία αυτή θα ευχαριστήσω την Ιστονική Προεδρία για την εξαιρετική δουλειά και τη συνεργασία της για τα θέματα αυτά. Εν τω μεταξύ, πραγματοποιήσαμε δεκάδες ώρες ωρών τρι, τριμερούς διαλόγου σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο και από την 1η Ιανουαρίου με την Βουλγαρική Προεδρία. η δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα είναι καλή. Καλύψαμε όλες τις διατάξεις που είναι κοινέ και για τις δύο προτάσεις και περιμένουμε ο πρώτος γύρος συζητήσεων για την πρόταση για τα σύνορα να ολοκληρωθεί την ερχόμενη εβδομάδα που συνολικά θα αφορά 60 άρθρα. Παραμένουμε με το τεράστιο έργο του ότι αν θέλουμε να συμφωνήσουμε επί ενός κειμένου ε, κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο και η Κομισιόν υποστηρίζουν και αυτές, ενδιαφέρουν και αυτοί για την επιτύχηση του στόχου. Όταν γίνεται μια μεταρρύθμιση, όλοι οι θεσμικοί παράγοντες πρέπει να είναι ανοιχτοί στην αλλαγή, τουλάχιστον εν μέρος, ενός μέρους της καθεστικής τάξης και να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις του Κοινοβουλίου. Άρα, ας είμαστε σαφείς. Δεν θα δεν θα υπερασπιστώ λιγότερο τις απόψεις του ε, Κοινοβουλίου μας ε, για προσχάρη μιας πρώτης συμφωνίας. Ελπίζω ότι η Κομισιόν θα είναι σωστός ενδιάμεσος ε, και θα προωθήσει το θέμα και ότι η Προεδρία θα είναι διατεθειμένη για συμβιβασμό όπως είναι και το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λένας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Για να συμπληρώσω, αυτά που είπε ο Κάρλος. Είναι ευπρόσδεκτος ο φάκελος για τις ε, ειδοποίησεις ε, επιστροφών του συστήματος πληροφοριών Σέγγεν. Για το θέμα αυτό έχουμε συνεργαστεί στενά με τους συναδέλφους της Επιτροπής. Καταλήξαμε σε ισχυρή κοινή θέση κατά την ψηφοφορία στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Το ανέφερε ήδη ο Κάρλος. Επανα Λαμβάνω, η συγκεκριμένη πρόταση βελτιώνει και επεκτείνει τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Σέγγεν, ώστε να είναι υποχρεωτικό για τα κράτη-μέλη να εισάγουν τις προειδοποίησεις στο σύστημα για αυτούς οι οποίοι έχει, ληφθεί απόφαση επιστροφής. Μια νέα κατηγορία ειδοποίησεων λοιπόν του συστήματος. Η θέση του Κοινοβουλίου είναι, λέει ότι είναι ευπρόσδεκτη η πρόταση και είναι χρήσιμο ειδοποίησεις να μπουν στο σύστημα και να χρησιμοποιηθούν για να επαληθεύσει η αναχώρηση των ανθρώπων αυτών οι οποίοι δεν έχουν τα προσόντα για διεθνή προστασία. Είναι σημαντικό η βελτίωση και είναι σημαντικό επίσης για τη θέση του Κοινοβουλίου τουλάχιστον είναι ότι αυτού του είδους οι ειδοποιήσεις δεν θα αλλάζουν τα δικαιώματα των προσφύγων ή των ετούντων άσυλο. Είναι μια λειτουργική βελτίωση και η αρχή των ρον ρεφουλμών, η θέση των ευάλωτων αντόπων ή παιδιών θα είναι απολύτως σεβαστές. Έχουμε τρεις πολιτικούς ε, τριμερείς διαλόγους με σημαντική πρόοδο, όχι πάντα τόσο ε, καλά όσο θα τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε και κάποια θέματα εξακολουθούν να εκκρεμούν και επίσης ε, αυτή που είναι αντικείμενο της ε, απόφασης επιστροφής ε, έχει προβλεφθεί εάν η εφαρμογή της απόφασης από το υπεύθυνο κράτος μέλος έχει εφαρμοστεί, έχει ανασταλεί ή έχει γίνει έφεση και εδώ έχουμε διαφορετικές απόψεις στον τριμερή διάλογο και συζητάμε πώς θα προσεγγιστεί το θέμα αυτό. Το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη η ταυτοποίηση να είναι όσο δυνατόν ακριβέστερη, χρησιμοποίηση δακτυλοσκόπησης και ε, φωτογραφιών Επίσης υπογραμμίστηκε στον τριμερή διάλογο ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν αυτόν όταν τα δεδομένα δεν είναι ε, διαθέσιμα, όταν ας πούμε η απόφαση για επιστροφή έχει ληφθεί ρήμην αλλά πρέπει εμείς να συνεχίσουμε να δίνουμε την έμφαση για την ακριβή ταυτοποίηση στην ακριβή ταυτοποίηση. Ένα, κάποια άλλα θέματα που συζητώνται σε τεχνικό επίπεδο και όπου είναι κάπως διστάμενες απόψεις προς το παρόν είναι η χρήση στατιστικών δεδομένων, τα άρθρα 6 και 11, η χρήση των ε, δακτυλικών αποτυπωμάτων σε σχέση με τις δακτυλοσκοπικές εικόνες της παλάμης, το θέμα της εισαγωγής και το θέμα των ειδοποιήσεων, η διαβουλεύση σε περίπτωση έβρεση των στοιχείων. Υπάρχουν διστάμενες απόψεις για αυτά. Προσπαθούμε να βρούμε ε, ε, συγκλίνωσες θέσεις και το θέμα του, στο, του σκοπού της επιστροφής. Ελπίζουμε και εδώ να σημειωθεί πρόοδο σύντομα. Με δύο λόγια. Πιστεύω ότι προκινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδης εισηγητές για την αφοσίωση, την επικοδομική συνεργασία και το πνεύμα συνεργασίας και πολλές ευχαριστίες προς το, τη Γραμματεία Κατρίν και όλους τους άλλους συμβούλους και βοηθούς. Κάναν πολύ καλή δουλειά πιστεύω ότι δουλεύουμε για την επίτευξη ενός θετικού αποτελέσματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα η Σκιώδης, ο κύριος Χαλάου, εκ μέρους των δύο άλλων, Ταμπίκ και Σίπλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το σύστημα πληροφοριών Schengen είναι σημαντικό σύστημα πληροφοριών που αντισταθμίζει την απουσία ε, ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Περισσότερο θεωρούμε ότι η ανάπτυξη του για την καλύτερη αντιμετώπιση μελλοντικών ε, απειλών είναι σημαντική. Ένας στόχος πρέπει να είναι η τεχνική αρχιτεκτονική του SIS με τρόπο ώστε να ενθαρρύνεται, ενισχύεται η αξιοπιστία του και να εξασφαλιστεί αδιάσπαστη ε, διαλειτουργικότητα του συστήματος. Θα πρέπει ε, αυτό να επιτευχθεί, παρότι σε εθνικό επίπεδο αυτό είναι θελοντικό. Εμείς θεωρούμε ότι το θέμα της τρομοκρατίας και της εσωτερικής ασφάλειας είναι σοβαρό και γι' αυτό θεωρούμε ότι η πρόταση να είναι υποχρεωτικές ειδοποίησεις για, ε, για τρομοκρατία δεν θα πρέπει να ενταχθεί στην αναλογικότητα. Αυτό αφορά την ασφάλεια των πολιτών. Επίσης, οι προϋποθέσεις για την έκδοση ειδοποίησεων για την είσοδο και παραμονή θα πρέπει να είναι ευέλικτες για να καλύπτονται οι ανάγκες των κρατών μελών. Η έκδοση μιας ειδοποίησης δεν θα πρέπει να συνδέεται με αυστηρά χρονικά περιθώρια ποινικών ποινών ε, όπως συμβεί μέχρι τώρα. Για να μην ενθαρρύνονται οι άτυποι μετανάστες να επανεμφανίζονται στα σύνορά μας θα πρέπει η αρχή αυτή της ειδοποίησης να ισχύσει γενικότερα. Θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα και στις περιπτώσεις που εμφανίζονται άνθρωποι στα σύνορά μας ισχυριζόμενοι ότι δεν έχουν ε, έγγραφα ταυτοποίησης. Τα βιομετρικά δεδομένα είναι λοιπόν σημαντικά. Καθώς η τεχνολογία για την ε, ε, επαλήθευση και την έρευνα με βιομετρικά συστήματα δεν εξελίσσεται, θα πρέπει να καθυστερήσουμε στη χρήση νέων εργαλείων. Όσον αφορά τι κατηγορίες δεδομένων που χρειάζονται για τι ειδοποίησει, η ανάγκη κάθε κατηγορίας θα πρέπει να μελετάται προσεκτικά, δεδομένου ότι υπερβολικέ Πολλέ πολλές πληροφορίες αποτελούν ε, διοικητικό άχθος και θόρυβο για το σύστημα. Η πρόσβαση στο SIS πρέπει να είναι αρκετά εκτεταμένη για να εξυπηρετούνται διάφοροι νόμιμοι, ε, νόμιμες ε, διαδικασίες. Όταν μιλάμε για προτάσεις επιστροφής, η πρόταση να γίνονται προσωρινά μη διαθέσιμες κάποιες ειδοποίησεις θα πρέπει να δούμε αν είναι εφικτό ή τεχνικά δυνατόν, τουλάχιστον να μην αποτελεί βάρος για κάποιους τελικούς χρήστες. Η πρόταση να μην εισάγονται ε, για τις εφέσεις κατά των ε, επιστροφών θα υπονομεύσει την όλη προσπάθεια. Το θέμα πρέπει να λυθεί, θα μπορούσε να λυθεί με, το, τη δημιουργία μιας ειδικής κατηγορίας για το αν είναι εκτελεστή ή όχι απόφαση όσον αφορά τη χρήση βιομετρικών δεδομένων για την αξιόπιστη ε, εντοπισμό ατόμων Είμαστε υπέρ της χρήσης ε, δακτυλοσκοπικών δεδομένων και δεδομένων ε, που αφορούν την εικόνα της παλάμης. Το δικαίωμα μετάδοσης δεδομένων για, σε τρίτες χώρες για τους σκοπούς της επιστροφής είναι σημαντικό για μια ε, αποτελεσματική και πιστική πολιτική επιστροφών. Οι υπερβολικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη μετάδοση μάλλον δεν θα έπρεπε να υπάρχουν υπερβολικές προϋποθέσεις για την μετάδοση αυτών των δεδομένων όταν μοναδικός σκοπός είναι να είναι πιο αποτελεσματικές επιστροφές. Τέλος, όσον αφορά τα πολιτικά θέματα που συζητώνται τώρα στα πλαίσια των τριμερούς διαλόγους, η ομάδα μας μπορεί να υποστηρίξει τους περισσότερους από τους προτινόμενους συμβιβασμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Μπέρκετ που μίλησε ονόματος κυρίας Μίριαμ Ντάλη Δυστυχώς η σκιώδη συγγήτρια συνάδελφος Ντάλι δεν μπορεί να παρευρεθεί. Θα σας διαβάσω τα σχόλιά της. Καταρχάς ευχαριστεί και τους δύο συγγητές και τους συνεργάτες τους για την ε, εντατική εργασία και την τόσο καλή συνεργασία το τελευταίο μήνα. Οι σοσιαλιστές και δημοκράτες υποστηρίζουν μέχρι στιγμής τις διαπραγματεύσεις για να ε, έχουμε ένα συμβιβασμό ε, μεταξύ της ασφάλειας και της ελευθερίας. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξακολουθήσει, να κρατάει τη γραμμή του ε, για κάποια ζητήματα κομβικής σημασίας. Και εδώ θέλω να σταθώ σε δύο συγκεκριμένα. Οι επιστροφές είναι απαράδεκτο για την ομάδα μας ε, να μπαίνει ειδοποίηση στο σύστημα SIS για μετανάστες που βρίσκονται εν μέσω της διαδικασίας προσφυγής. Ε, δεν έχουν εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα και αν επιτρέπει ε, η διαδικασία και η νομοθεσία να τις χρησιμοποιήσουν, θα πρέπει να τους αφήνουμε να τις χρησιμοποιήσουν. Παρ' όλα αυτά το Συμβούλιο διαφωνεί. Ως συμβιβασμό πρότεινε ο εισηγητή στο πάγωμα ή, ε, να μην φαίνεται ειδοποίηση, αλλά ούτε αυτό αρέσει στο Συμβούλιο και θυμίζω και στον κύριο Λένας ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη η θέση του Κοινοβουλίου ε, για την διαδικασία και τον υποστηρίζουμε. Για τα άλλα δύο θέματα οι διαπραγματεύσεις ήταν καλές, ωστόσο έχουμε ε, να αντιμετωπίσουμε τεράστια κρίση. Ε, αν, ε, πρέπει να κρίνουμε ποια στοιχεία θα μπουν. αυτό το κατόφλι είναι χαμηλότερο από εκείνο που προβλέπει το Ευρωπαϊκό Ένταλμα και οι ορισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σοβαρό έγκλημα. Η δική μου πολιτική ομάδα ανέκαθεν ήταν υπέρ της τριετίας, αλλά η ε, Επιτροπή αποφάσισε ε, η δική μας να υποστηρίξει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει να το σεβαστούμε. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε προς τον κύριο Κοέγιο και το Συμβούλιο ότι η σημερινή πρόταση του Συμβουλίου που καλεί τα κράτη-μέλη να, ε, δώσουν, να έχουν λευκή επιταγή για το ποιον θα εισαγάγουν στο σύστημα είναι απαράδεκτη με οποιαδήποτε μορφή τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι ε, σωρεύουμε ε, στοιχεία για παραβάσεις, για τη μικροπαραβατικότητα, για κλήσεις της τροχέας και πάει λέγοντας. Δεν είναι αυτό οργανωσμένο έγκλημα, τρομοκρατία ή σοβαρό έγκλημα. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στην Επιτροπή μας γι' αυτό. Δεν έχουμε συμφωνήσει και σας παρακαλώ στην μελλοντική συνάντηση του τριμερούς διαλόγου να ληφθεί υπόψη αυτό. Θέλουν το λόγο άλλα μέλη. Όχι. Ε, δεν ξέρω, οι συγητές θέλουν να απαντήσουν. Ο κύριος Κοέγιο. Ευχαριστώ. Δύο λόγια. Για το τελευταίο αυτό σημείο. Συμφωνώ με την άποψή σου Νομίζω ότι πρέπει να παραμείνουμε στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά θα πρέπει να αξιολογήσουμε τι θέλουμε να προστατεύσουμε τελικά. Σε ό,τι αφορά την εισαγωγή ε, προειδοποίησεων, ή ειδοποίησεων καλύτερα, ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα, ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από κράτος σε κράτος. Νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναδούμε τα πράγματα. Γιατί αν δεν εναρμονίσουμε τα πράγματα με κάποιο τρόπο, τελικά το κάθε κράτο μέλο θα αντιμετωπίσει τελείω διαφορετικά τι ειδοποίησει. Ε, ποιο είναι το status quo τώρα, ότι είναι θέμα εθνική αρμοδιότητα. Επομένω, οποιαδήποτε βήματα μπορούμε να πάρουμε, ούτω ώστε να βάλουμε ένα κάποιο επίπεδο εναρμόνισης θα είναι θετικό. Φυσικά, πολιτικά, θα πρέπει να δούμε σε επίπεδο Ευρώπης εάν τελικά η πρόοδος μας ικανοποιεί. Φυσικά θα πρέπει να φτάσουμε σε συμβάσμα όμω για κάτι τέτοιο με το Κοινοβούλιο και ελπίζω ότι η Βουλγαρική Προεδρία θα παροτρύνει και θα δώσει έτσι ε, κίνητρα στο Συμβούλιο τόσο ώστε να φτάσει σε μια θέση που θα, το επιτρέψει, θα το επιτρέψει να συμβαστεί μαζί μας. Ίσως τελικά η τελική λύση δεν θα είναι πολύ κοντά στην ισχυρή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν θα είναι τόσο ούτε όμως εκεί που βρίσκεται το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Κάπου στη μέση. Για να δούμε λοιπόν ποιο θα είναι το μέλλον των διαπραγματεύσεων και τι θα δώσουν, τι καρπούς θα δώσουν. Ευχαριστώ Κάρλος. Πολύ ωραία. Υπάρχει τώρα η συνεδρίαση της κοινή Επιτροπής ε, μαζί με την Επιτροπή Γυναικών. Θα πρέπει να περάσουμε στην αίθουσα 3E2. ε 2 Σας ευχαριστώ.